Η Οι αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μας γνωστοποίησαν την εκλογή του κ. Ντάνιελ Ντόρτον για να αντικαταστήσει τον κ. Φίλιπ Μπράντμπορν από τις 8 Ιανουαρίου και μετά. Και σύμφωνα με τα ισχύοντα, ο κανονισμός προβλέπει ότι από τις 8 Ιανουαρίου και μετά εκλέγεται και επίσημα ο συνάδελφος τον καλωσορίζω και του τονίζω ότι μέχρι να ε, δοθεί η έγκριση των διαπιστευτηρίων του θα μπορεί να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων του εφόσον έχει υπογράψει την προβλεπόμενη δήλωση συμφερόντων. Και τώρα περνάμε στις ψηφοφορίες.